Σύμφωνα με το άρθρο 219 παράγραφος 2 του κανονισμού, οι υποψήφοι ή υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν μια σειρά συγκεκριμένων όρων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μόνο τις όρους εκείνους που μας αφορούν άμεσα, σας αφορούν άμεσα. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει προταθεί από τουλάχιστον 40 μέλη, από τουλάχιστον 2 κράτη-μέλη. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζει κανείς ε, περισσότερο από έναν υποψήφιο ταυτόχρονα. Σε περίπτωση που ένας βουλευτής ε, υποστηρίξει πιο πολλές υποψηφιότητες με την υπογραφή του, δεν θα ισχύσει καμία από τις υπογραφές αυτές. Αυτό στην περίπτωση, ε, χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε την υποψηφιότητα του εκάστοτε ατόμου. Και όταν λοιπόν αν έχετε λοιπόν αποφασίσει και μόλις λάβω την υπογραφή σας, δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η υπογραφή. Σύμφωνα με το 19 παραγραφός 3 του κανονισμού, θα ε, διαβιβάσω όλες τις υποψηφιότητες που πληρώνουν τους απαραίτητους όρου στην Επιτροπή ε, α, Και αυτή η λίστα λοιπόν θα η Επιτροπή θα διοργανώσει ακροάσεις το Δεκέμβριο, οι οποίες θα είναι ανοιχτές σε όλους. Η εκλογή λοιπόν θα γίνει τον Ιανουάριο του 2015 και οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης της Προεδρίας φυσικά είναι στην διάθεσή σα για οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση έχετε. Οι αρμόδιες ε, Επιτροπής ε, έχουν ε, υποβάλει κάποια διευθυντικά σε πέντε κείμενα που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 2331 θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά αυτά εκτός και αν υπάρχει ένταση μέσα, μέσα 24 ώρες και τα έχετε λοιπόν τα διευθυντικά αυτά στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας θα δημοσιευθούν και στα πρακτικά της συνεδρίασης